για νομοθεσία, νομοθετικό έργο στο μέλλον. Πρέπει αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα με μια λύση που θα ικανοποιήσει όλου. Η κυρία Παπαδοπούλου. Πρόεδρε, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η